Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen. Κυρίες και κύριοι, λοιπόν, πάμε στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια. Η Εισηγητής ο κύριος Σαουντάργας. Ψηφίζουμε το σχέδιο έκθεσης. Έχετε στα χέρια σας το κατάλογο ψηφοφορίας κανονικά και είχατε και την ευκαιρία να αναπαυθείτε. Αρχίσαμε στις 10 η ώρα. Εσείς μια χαρά ήρθατε, όχι όλοι μας βέβαια γιατί οι συντονιστές ήρθαν από τις 9. Λοιπόν, ε, ψηφίζουμε. Αγαπητοί φίλοι, ψηφίζουμε δοκιμαστικά πρώτα, όπως ξέρετε. Σας αρέσει η Επιτροπή Ήτρε, ψηφίστε παρακαλώ, ηλεκτρονικά. Άρχεται η επαλήθευση. Ψηφίσατε. Κάνουμε ένα ηλεκτρονικό έλεγχο. Πέρας. Α, καλά τα πάμε. Έχουμε και κατά, έχουμε και αποχές κάθε φορά θα ελέγχουμε την αποδοχή αν αυξάνεται ή αμειώνεται το μεδόν. Πότε είναι οι επόμενες εκλογές, α, σε τέσσερα χρόνια. Έχουμε χρόνο πολύ. Αλλά δεν πειράζει να φροντίσουμε να αυξηθεί η αποδοχή μας. Όλα, όλα είναι προεκλογική εκστρατεία, ό,τι και να κάνεις. Α, κατά τα άλλα έχουμε κανένα Βρετανό παρόντα σήμερα εδώ. Ποιος είναι από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, συνεργάτες βοηθεί ίσως. Καλή τύχη σε όλους. Καλή τύχη, τίποτα άλλο. Καλή επιτυχία. Λοιπόν, σχόλια ακούγονται από κάτω, δεν τα ακούμε εμείς. Αγαπητοί συνάδελφοι, αρχίζουμε. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο και θα είναι μακρά η ψηφοφορία, πολύ. Compromise Amendment Συμβεβαστική 1 είπε κατά άποχες εγκρίνεται. 131 τροπολογία ψήφι υπέρ κατά η ηλεκτρονική υπολήθευση αρχίζει για την 131. Πέρας. απορρίφτεται. Η συμβιβαστική υπαριθμό 2. Ψηφίπε. Κατά αποχές εγκρίνεται. 135. είπε. Κατά. Αποχές πρέπει να το ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Η συμβιβαστική 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 220 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 164 υπέρ. Κατά. Πρέπει να το ελέγξουμε. Αρχίζει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίψετε. Η συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. Η συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Απόχες Εγκρίνεται. Η 192 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 197 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 200 ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 201 υπέρ, κατά, Νομίζω ότι έχει εγκριθεί, αλλά το ελέγξουμε. Άρχεται η σφοφόρια 201. Πέρας. Εγκρίνεται. 202 υπέρ. Κατά. Αποχές. Μάλλον έχει εγκριθεί. 203 υπέρ. Against Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 208 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η συμβαστική 7 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 223 υπέρ, κατά. Ε, παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Η 223 είναι. Πέρας. Rejected. Απορρίπτεται. 2.21 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ή 11 το πρώτο τμήμα ψήφι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 8 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 16 είπε. κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 9 είπε. κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 10 διότι 253 εξ όσων γνωρίζω έχει αποσυρθεί. Σωστά τα λέω. Ωραία. Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 272 υπέρ κατά έλεγχος ζητώ συγγνώμη πέρας εγκρίνεται η 270 υπέρ κατά μάλλον χρειάζεται και πάλι έλεγχο αρχίζει η ψηφοφορία λίγη εγκρίνεται. Ζητώ συγγνώμη. Η 11 συμβιβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 282 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 286 υπέρ κατά Ζητώ συγγνώμη, αλλά θα πρέπει να την ελέγξουμε. 286 ηλεκτρονική υπαρήθευση. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 294 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Η 13 είναι η συμβιβαστική υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Η 313 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ για την τροπολογία 313. την ψηφοφορια ψηφοφορία, πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 13α, ψηφι π. υπέρ. 13α υπέ. Κατά. Αποχές πρέπει να ελέγξουμε. Η Ηλεκτρονική επαλήθευση λοιπόν. Να έρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Η τροπολογία υπαριθμών. Όχι εννέα. Τι έγινε η 342. Ε, την εννέα θα ψηφίσουμε υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι έχει απορριφθεί αλλά χρειάζεται έλεγχο εννέα. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 11 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Επίσης απορρίπτεται. Έλεγχος. Ελέγχουμε την 11 ηλεκτρονικά. Closed. Accepted accepted. So we go to 314. Uh, uh, Πάμε στο 314. 314. Πρώτο τμήμα. 314 το πρώτο τμήμα ψηφίζουμε. Ψηφί υπέρ παρακαλώ. Κατά. Άποχες. Έλεγχος παρακαλώ και πάλι γιατί 314 αρχίζει τώρα. Και μάλιστα το πρώτο τμήμα. Πέρας. Απορρίπτεται. Τώρα πάμε στην 319 πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται αυτή τη φορά. Θέλετε έλεγχο. Ωραία. Να την ελέγξουμε. 319 το πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία πέρας. Accepted. So we go... Εγκρίνεται. Είναι πάρα πολύ μακρύς ο κατάλογος. Πάμε στη 3.14 μέχρι και την 3.40 μαζί. Είναι μαζί και η 3.19, 3.39 κλπ. Γιατί είναι ταυτόσιμες. Τέσσερις τροπολογίες μαζί θα ψηφίσουμε. Ψήφιπε. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αλλά ας το ελέγξουμε καλύτερα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα. Άρχεται η ψηφοφορία. Closed. Πέρας. Εγκρίθηκε. Λοιπόν, άρα θα πάμε τώρα στο επόμενο μπλοκ τροπολογιών 3.14-3.19 ε, ταυτίζονται αυτές οι δύο και θα τις ψηφίσουμε μαζί. Ψήφι κατά απόχες εγκρίνεται. Τρία δεκαεννιά, τώρα το δεύτερο τμήμα, μαζί με την 3.21 θα ψηφίσουμε. Και αυτές είναι ταυτόσιμες. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 3.15 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Η συμβαστική 14 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Η 3.43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3.41 υπέρ. Κατά. Άποχες. Έλεγχος για τη 3.41 παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία και τελειώνει. Εγκρίνεται. 3.47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3.45 υπέρ. Α, συγγνώμη, μαζί με την 346 είναι η υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίπτεται. Okay, check. Α, έλεγχο θέλετε, ωραία. Και τις δύο πάλι μαζί. Καλή ιδέα να τσακάρουμε καμιά φορά. 3.45 και 3.46. Άρχεται και λίγη αμέσως. Απορρίπτεται αυτή τη φορά. Κατά τύχη το είχα πει σωστά. Συμβαστική 16 πέ. Κατά άβοχες εγκρίνεται. Η 351 το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Παρακαλώ. 351 το δεύτερο μέρος. Άρχη ψηφοφορία. Λίγη. Εγκρίνεται. 348 υπέρ. Κατά απόχες εγκρίνεται. 3,70 υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται. Η συμβιβαστική 17 υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται. 3,74 η τελευταία πρόταση. Τελευταία πρόταση μόνο υπέρ. Against. Κατά. Άποχες. Έλεγχος. Open. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Τρία, επτά, οκτώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3,79 υπέρ. Κατά. Αποχές. Αποδεκτή. Συμβαστική 18 υπέρ. Κατά αποχές αποδεκτή 386 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε ελέγχουμε ηλεκτρονικά 386 άρχεται πέρας αποδεκτή Δύο μαζί η 366-415 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε τις δύο προπολογίες, 366 και 415. Άρχεται η ψηφοφορία. Κλείνει. Απορρίπτεται. Ισοψηφία. Γι' αυτό πρέπει να ελέγχουμε συχνά. 394 υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε παρακαλώ. 394 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Το ίδιο αποτέλεσμα απορρίπτεται. 37 υπέρ. Κατά αποχές. Ελέγχουμε, αν δεν το είχατε καταλάβει. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Βλέπετε, εγκρίνεται. Ένα λεπτό. Έντεκα. 313 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε παρακαλώ. 413 ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία πέρας. Απορρίπτεται αυτή τη φορά. Συμβαστική 19 υπέρ. Κατά. αποχές μάλλον γίνεται αποδεκτή, αλλά ας ελέγξουμε. Συμβιβαστική 19, ας ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρας. Εγκρίνεται. 405 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 408 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 408. εφόσον επιθυμείτε θα ελέγξουμε, άρχεται η ψηφοφορία, πέρας, απορρίπτεται. 369 υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίφθηκε. Απορρίπτεται, συνάδελφοι. Θέλετε να ελέγξουμε, ελέγχουμε. 369, έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Α, αποδεκτή. Εγκρίνεται. Ποτέ δεν αρνούμε ελέγχους. Γιατί δεν σηκώνετε τα χέρια σωστά δεν τα βλέπω. Σας ευχαριστώ. Συγχαρητήρια κυρία μου. Εξαιρετική ιδέα σας. 417 υπέρ. Κατά. Αποχές. Αποδεκτή. 418 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε την 418. 418 έλεγχος. Πέρας. Απορρίφθηκε. 416, 316 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε παρακαλώ να σηκώνετε τα χέρια ευκρινώς. 416. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται. Είναι αδύνατο να κάνω σωστή καταμέτρηση έτσι. 421 υπέρ. Κατά. Αποχές αποδεκτή. 414 υπέρ. Κατά. Αποχές ας ελέγξουμε. Πρέπει να ελέγξουμε. Άρχεται και πέρασε. Απορρίπτεται. 367 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε παρακαλώ. 367 έλεγχος. Πέρας. Αποδεκτή. Συμβιβαστική 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Αποδεκτή. 480 υπέρ. Κατά. Αποχές αποδεκτή. 419 υπέρ. Κατά αποχές αποδεκτή. Συμβιβαστική 20α υπέρ. Κατά αποχές αποδεκτή. 445 υπέρ. Κατά αποχές αποδεκτή. 443 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 450 υπέρ. Κατά αποχές αποδεκτή. 451 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 452 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 453 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε. 453 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. 454 υπέρ. Κατά. Αποχές. Αποδεκτή. Με την ίδια πλειοψηφία συμβαστική 20B υπέρ. Κατά. Αποχές αποδεκτή. Συμβαστική 21 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική. 252 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 22 υπέρ, κατά αποχές αποδεκτή 31 υπέρ, κατά αποχές αποδεκτή 478 υπέρ, κατά αποχές αποδεκτή 482 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 448 υπέρ, κατά ας ελέγξουμε. Με συγχωρείτε 483. Ελέγχουμε. 483. 483. Πέρας. Αποδεκτή. Παρακαλώ να σηκώνετε τα χέρια σας. 484 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 485 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε παρακαλώ. 485 έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Αποδεκτή. 486 υπέρ. Κατά. Αποχές ίδια πλειοψηφία. Εγκρίνεται. 487 υπέρ. Κατά. Δεν είναι σαφές. 487 ελέγχουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος παρακαλώ. 38. Πέρας. Εγκρίνεται. 191 υπέρ. Κατά. 491. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα πρέπει να ελέγξουμε την 491. Ελέγχουμε παρακαλώ. Πέρες. Εγκρίνεται. 365 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 23 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 516 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 505 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 504 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 24 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 507 υπέρ, κατά αποχές αποδεκτή. 506 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 25 υπέρ, κατά αποχές αποδεκτή. 535 υπέρ, κατά αποχές ας ελέγξουμε παρακαλώ ...535 ηλεκτρονικός έλεγχος... ...πέρας... ...εγκρίνεται... ...534 υπέρ... ...κατά αποχές θα πρέπει να ελέγξουμε 534 έλεγχος. Πέρας. Εγκρίνεται. 606 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 26 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 27 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 166 υπέρ. Κατά αποχές αποδεκτή. Συμβασμός 28 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 29 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 571 υπέρ. Κατά Ας ελέγξουμε παρακαλώ. 571. Έλεγχος. Πέρας. Εγκρίνεται. Με μικρή πλειοψηφία. 586. Πέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αποσύρεται η 583 584 υπέρ. Κατά. Αποχές αποδεκτή. 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 589 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 590 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 588 υπέρ. Κατά. Πρέπει να ελέγξουμε. 588 ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίπτεται. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές αποδεκτή συμβιβασμός 30 υπέρ. Κατά. Αποχές αποδεκτή. 603 υπέρ. Κατά. Θα πρέπει να ελέγξουμε. 603. Άρχεται ο έλεγχος. Πέρας. Αποδεκτή. 604. Υπέρ. Κατά. Αποχές Ας ελέγξουμε. Ελέγχουμε. 604. 604. Πέρας. Απορρίπτεται. 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Αποδεκτή. 659 υπέρ. Κατά. Αποχές αποδεκτή. 605 υπέρ. Κατά. Αποχές αποδεκτή. 635 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 31 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 608 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ωραία, ελέγχουμε. 608. 608 πέρασε. Απορρίπτεται. Με μικρή διαφορά. 662 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 615 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 32 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 32α υπέρ. Κατά αποχές αποδεκτή 631 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 633 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 634 υπέρ. Κατά αποχές αποδεκτή. Θέλετε να ναι. ελέγξουμε. Εγώ είπα ότι έγινε αποδεκτή. Εντάξει, εντάξει, αστείαφομαι. Άρχεται η ψηφοφορία. Είμαι ανοιχτό σε κάθε πρόταση. Θα δούμε, θα δούμε. Αλλά ψηφίστε, σας παρακαλώ. Είδατε που εγκρίθηκε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί ήταν ε, δική μου η τροπολογία φαίνεται ότι αλλάξατε γνώμη, δεν ήταν απόλυτα σαφές. Συμβαστική 34 υπέρ. Κατά αποχές ε, αποδεκτή. 636 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Εντάξει, εντάξει, ελέγχουμε. Πολύ καλή ιδέα. 6.36 ελέγχουμε. Πέρας. Η ισοψηφία, άρα απορρίπτεται. Αλλά είχατε δίκιο ότι έπρεπε να γίνει έλεγχος. Δεν ήμουν απόλυτα βέβαιος. 475 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε. Πέρας. Αποδεκτή. 630 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε, ας ελέγξουμε και πάλι. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 34α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 646 υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται. 647 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 648 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 35 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 35α υπερκατά, αποχές αποδεκτή. Συμβαστική 36 υπέρ. Κατά αποχές αποδεκτή. 36α υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 37 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 688 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, ε, ελέγχουμε. 688. Έλεγχος. Πέρας. Απορρίπτεται. 689 υπέρ. Κατά. Αποχές. Αποδεκτή. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Αποδεκτή συμβιβαστική. 10. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Όχι. Με συγχωρείτε, λάθο λάθος. Συμβιβαστική 38α. Υπέρ. Κατά. Πρέπει να γίνει έλεγχος. Αρχίζει η ψηφοφορία. Επί της 38α. Πέρας. Αποδεκτή. Δέκα πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές ε, εγκρίνεται. τρία υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. τέσσερα υπέρ. Κατά. Αποχές Ας ελέγξουμε. Είναι τα τέσσερα Ελέγχουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Είναι τα 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 760 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Είναι τα 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 181 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 698 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 701 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 700 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε. 700 έλεγχος. Πέρας. Απορρίπτεται. 699 υπέρ. Κατά. Αποχές. Πρέπει να ελέγξουμε. Σας παρακαλώ να σηκώνετε τα χέρια γιατί δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. 699 ελέγχουμε. Πέρας. Αποδεκτή. 704 υπέρ κατά αποχές πρέπει να ελέγξουμε γιατί μεγάλη αποχή 704 ελέγχουμε πέρας απορρίπτεται 702 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 703 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 703 απορρίπτεται. Θέλετε έλεγχο? Ωραία, ελέγχουμε. 703. 703. Πέρας. Απορρίπτεται. 705. Υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε. 705 έλεγχος. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 39α υπέρ. Κατά. Αποχές ε, εγκρίνεται. 737 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 40α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 40β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 739 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 40γ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβιβαστική 41. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 748 υπέρ, κατά, αποχές. Ας ελέγξουμε, ας ελέγξουμε. 748. 748 αρχίζει ο έλεγχος. Πέρας. Απορρίπτεται. 25 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 762 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 753 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 754 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά Ας ελέγξουμε, ας ελέγξουμε. Μάλλον γίνεται αποδεκτή. Ελέγχουμε τη 12 ίντα. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 43 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 761 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 685 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 769 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 43α υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 778 κατά αποχής απορρίπτεται 776 υπέρ κατά πιθανότατα εγκρίνεται αλλά ας ελέγξουμε 776 έλεγχος παρακαλώ 776 επαναλαμβάνει ο πρόεδρος Πέρα του ελέγχου Εγκρίνεται. 779 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 781 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε. 781. Πέρας του ελέγχου. 777 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 799 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ας ελέγξουμε. 799 έλεγχος. Πέρας του ελέγχου. Απορρίπτεται. Έκπληξη. 798 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. στο το ελέγχου. Εγκρίνεται. 808 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 801 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 802 και 807 από κοινού. Ταυτόσιμες. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. Είναι τα 15. Δεύτερο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Είναι τα 15 δεύτερο μέρος έλεγχος. Έλεγχος. Πέρας του έλεγχου. Απορρίπτεται. 803 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 805 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 806 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 804 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Είναι τα 13 υπέρ, κατά, αποχές, αποδεκτή. 759 υπέρ, Όχι, λέει ο πρόεδρο. Αυτή είχε, γίνει, είχε εγκριθεί. Ένα λεπτό. Συμβιβαστική 49 λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 812. 812. Υπέρ. 812 υπέρ. Μιλούμε για την 812 κατά. Αποχές πρέπει να ελέγξουμε λέει ο πρόεδρος. Έλεγχος για την 812. Μάλλον απερίφθη, αλλά το ελέγχουμε. Το ελέγχουμε. Πέρα στο ελέγχου. 815 υπέρ κατά αποχές 8.16 8-16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8-20 υπέρ κατά αποχές εγκρινεται 8.19 8-19 υπέρ κατά αποχές έλεγχος έλεγχος για την 8-19 Πέρας του έλεγχου. Απορρίπτεται. 818 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 821 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε. Έλεγχος 821. πέρας του ελέγχου ε, εγκρίνεται. Ε, συμβαστική α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ κατά αποχές Λοιπόν, να ελέγξουμε λόγω μεγάλου αριθμού αποχών. 42 έλεγχος. Πέρασε. Ναι, όχι, απορρίπτεται. 40. Υπέρ, κατά, αποχές. Ελέγχουμε. Ελέγχουμε. Πέρασε εγκρίνεται. Συμβαστική D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. F α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 62 υπέρ κατά να το ελέγξουμε ελέγχουμε στο 62 Ελέγχουμε. Πέρα στο ελέγχου. Απορρίπτεται. 63. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος, έλεγχος. 63 έλεγχος. Closed. Rejected. Rejected. Compromise I in favor. Συμβαστική γιώτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 122 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 70 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε την, την 70, ελέγχουμε την 70 πέρας του ελέγχου εγκρίνεται. 77 υπέρ κατά αποχής εγκρίνεται. 120 υπέρ υπέρ κατά αποχής εγκρίνεται. Όχι, ας ελέγξουμε. Ας ελέγξουμε. 120. 120 έλεγχος. Πέρας. Εγκρίνεται. 79 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 94 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 90 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική L υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 102 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 69 υπέρ. Κατά αποχές να την ελέγξουμε την 69. 69. Πέρα του ελέγχου. Εγκρίνεται. 85 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ας την ελέγξουμε. Ελέγχουμε την 85. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβαστική αίμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 100. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 68. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 93 υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται. 104 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 103 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 105 υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται. 106 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 124 υπέρ κατά αποχές ας την ελέγξουμε έλεγχο στην 124 πέρας εγκρίνεται συμβαστική όμικρον υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται 125 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 123 υπέρ κατά αποχές ας το ελέγξουμε. Έλεγχο στην 123 παρακαλώ. Και πέρα στο ελέγχου. Εγκρίνεται. 118 υπέρ. Κατά. Αποχές Ας την ελέγξουμε. Ελέγχουμε την 118 ηλεκτρονικά. Πέρας. Εγκρίνεται. 121 υπέρ. Κατά. Εποχές. Αποδεκτή. 119 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Έλεγχος στην 119. Πέρας. Απορρίπτεται. Um, uh, uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε ένα, μια πρόταση του εισηγητή για τις ε, παραθέσεις, για τις παραπομπές, να ψηφίσουμε en Εάν κάποιος αρνείται, τότε θα πρέπει να πάμε τροπολογία προς τροπολογία. Πρέπει να έχουμε ομόφωνη συμφωνία σε αυτό. Πατήστε το κουμπί σας και πείτε ναι, όχι. Διαφωνείτε λοιπόν. Ναι, Πρόεδρε. Διαφωνώ. Μάλιστα. Επομένως μία προς μία. Αγαπητοί φίλοι, είναι εκπαίδευση για την επόμενη ψηφοφορία. Λοιπόν, 3, 1, 17, 18 και 19. Εδώ πρέπει να ψηφίσουμε μαζί γιατί είναι ταυτόσιμες. Μαζί με την 3. Όχι, όχι. Πρώτα η 3. Πρώτα η 3 μόνη της. 3.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 και κάποιοι συνάδελφοι ήταν ε, κατά ορισμένων τροπολογιών, επομένως ήταν σημαντικό να τις ε, ελέγξουμε. Σα ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Και πάμε τώρα στην ηλεκτρονική ονομαστική ψηφοφορία για το σύνολο της προτάσεως. Παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Παρακαλώ συνάδελφοι να το προσέξουμε λίγο εδώ αυτό. Έχετε ψηφίσει πέρας της ψηφοφορίας. 42 υπέρ 13 κατά 4 αποχές συγχαρητήρια στον κύριο εισηγητή. Εάν ε, θέλετε ο κύριος εισηγητή θα ήθελε κάτι να μας πει. Ο κύριος Ταουντάρκας παρακαλώ να ευχαριστήσω όλους για την πολύ σκληρή δουλειά και ευχαριστώ όλους για την υποστήριξη. Ευχαριστώ λέει και ο Πρόεδρος. Hello. Colleagues, let's continue. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε. Ο κύριος Μπούζεκ χρειάστηκε να αποχωρήσει για μια σημαντική συνεδρίαση στην Πολωνία και μου ζήτησε να τον αντικαταστήσω. about the work of the Λοιπόν, το έργο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς, ΕΝΤΣΟ, στο πλαίσιο της Ενεργειακής Ένωσης θα χαρούμε μία παρουσίαση από την οργάνωση αυτή και θα ανταλλάξουμε απόψεις στη συνέχεια. Θα ήθελα πάρα πολύ να καλωσορίσω την κυρία Βέντε Χάγεν που είναι αντιπρόεδρος ε, για την Ευρώπη και τον κύριο Βιτόριο Μπουσάτσι όπου είναι ε, ο Γενικός Διευθυντής ε, του G. Τι είναι αυτό, είναι για το φυσικό αέριο. Thank you. <clears throat> That ENSO for European... σε θυμίζω, είναι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς. Το ε δηλαδή είναι ε, ε, δεξισμός δεν είναι Ευρώπη και το G είναι gas, δηλαδή φυσικό αέριο. Για να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ ε, διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς στην Ευρώπη για να εξασφαλίσουμε την ανάπτυξη ενός συστήματος πανευρωπαϊκού ευθυγραμμισμένο με τους στόχους ε, τους ενεργειακούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλό θα ήταν να κάνετε λίγη ησυχία. Λοιπόν, έχουν οριστεί από το τρίτο πακέτο ε, της ενεργειακής αγοράς το 2009 και έχουν λάβει και αντίστοιχη εντολή για την περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς ε, ηλεκτρισμού και ε, φυσικού αερίου. Έχουμε ένα τέταρτο το και μία ώρα ε, για να ε, δούμε αυτό το θέμα, ίσως να μην την εξαντλήσουμε. Θα δώσω το λόγο πρώτα στην κυρία Χάγκεμ. Έχετε ακριβώς 7 λεπτά ή και λιγότερο αν δεν χρειάζεται να τα εξαντλήσετε. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Λέγομαι Μπέντε Χάγκεμ, είναι αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΝΣΟΗ και έχω εκλεγεί και πρόεδρος για την επόμενη διετία. Ξέρετε ποια είμαι λοιπόν τώρα. Πώς συνεισφέρουμε εμείς και τι πρέπει να κάνουμε να εξασφαλίσουμε τον εφοδιασμό, τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια όλων αυτών. The energy trilemma. Έχουμε ένα τρίλημα στην ενέργεια και είναι ένας στόχος πάρα πολύ δύσκολος θα πρέπει να έχουμε πολιτικές που θα ε, πρέπει να λύσουν αυτό το τρίλημα και αυτό είναι ε, μία από τις πιο δύσκολες προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν κυβερνήσεις και ε, οικονομία. Η Ενεργειακή Ένωση δημιουργήθηκε για να λυθεί αυτό το ενεργειακό τρίλημα και οι TSOs που είναι οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς είναι κρίσιμος παράγων, το γνωρίζουμε και θέλουμε και εμείς να συνεισφέρουμε για να βοηθήσουμε με αυτό το σημαντικό έργο και εργαλείο. Θα ήθελα λίγο να θυμίσω ποια είναι η επίσημη εντολή μας. Είναι το τρίτο αυτό ενεργειακό πακέτο περί του οποίου πρόκειται οδηγία για το ηλεκτρικό ρεύμα και για το φυσικό αέριο. ENSO-E, ENSO-G και ACER. Αυτά είναι τα εργαλεία που έχουμε και τα μέσα στη διάθεσή μας. για να γίνει ε, απρόσκοπτα αυτή η ενεργειακή μετάβαση. Hmm. This is very delicate. Πολύ ευαίσθητο αυτό το μηχάνημα. Serving 41, uh... 34 χώρες έχουμε 41 συστήματα ε, που είναι όλα εθνικά μονοπόλια και οι διαχειριστές και οι ρυθμιστές ε, ενέχονται σε αυτή την προσπάθεια. Έχουμε 1000 ε, γίγαβατ στην παραγωγή στην Ευρώπη και 30.000 χιλιόμετρα συνδέσεων, καλωδίων. Ποιοι είναι οι βασικοί μας στόχοι. Να αναπτύξουμε ένα πρόγραμμα Δέκα ετές. Θα επανέλθω σε αυτό. Και επίσης ε, ένα κώδικα ε, νομοθεσία πάρα πολύ λεπτομερή για την διευθέτηση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Δημιουργούμε νέες αγορές και συνεργαζόμαστε σε περιφερειακό επίπεδο. Επίσης πολύ σημαντικό αυτό για μας, η περιφερειακή συνεργασία. Εκτός από την ευρωπαϊκή. Και είμαστε και σύμβουλοι πολιτικής σε διάφορα θέματα των αρμοδιοτήτων μας. Επενδύουμε 150 δισεκατομμύρια ευρώ στην ευρωπαϊκή υποδομή ε, με ορίζοντα 2030 είναι μόλις το 1 τρίτο των συνολικών επενδύσεων στην Ευρώπη. Και αν δούμε το πακέτο Juncker, ε, τελικά θα είναι πολύ περισσότερα αυτά. Πρόκειται για μεγάλη επένδυση και την ώρα που συζητούμε εδώ εμείς επενδύουμε. 25.000 ε, χιλιόμετρα ε, ε, ρεύματος σταθερού και 30.000 είναι μεταλλασσόμενο. 60% της συνολικής κατανάλωσης καλύφθηκε και θα μειωθεί η τιμή από 2 μέχρι 5 ευρώ ένα μεγαβατ ώρα. Δηλαδή, χοντρικά, ε, ε, εάν ε, επενδύσουμε εμείς στην Ευρώπη, το κέρδος από ένα ευρώ που θα επενδυθεί είναι δύο ευρώ. Χρειαζόμαστε λοιπόν και κανονισμούς και έχουμε κώδικες ε, τρεις για τον ηλεκτρισμό, τρεις για την ε, σύνδεση στο δίκτυο και τέσσερις για τη λειτουργία. Είναι χίλιες, χιλιάδες σελίδες κανονισμών που θα εγκριθούν το 2015. για να γίνει η αγορά ενέργειας επιτυχία. Δεν κάνουμε μόνο κανονισμούς όμως. χτίζουμε και νέες αγορές. Και έχουμε τη μεγαλύτερη πολυεθνική αγορά ενέργειας στον κόσμο. Κάνουμε ε, πληστηριασμούς για 23 συστήματα με τεράστιες ε, ωφέλειες. Πέφτουν οι τιμές, πέφτουν οι εκπομπές και ε, βελτιώνεται η διαχείριση και η λειτουργία καθώς επίσης και η ασφάλεια του συστήματος. Στις 15 Μαΐου πέρσι ε, ήταν ίδια τιμή στη θάλασσα του Μπάνιτς και στην ε, Χερσόνησο. Και το 2015 η Τσεχική Δημοκρατία, ε, η Ρουμανία, η, η η ε, Ουγγαρία και η Σλοβακία θα μπουν στην αγορά. Και έχουμε και θα, έχουμε την ίδια τιμή στην ε, Μαύρη Θάλασσα. Και αυτό όλα για συνεχές και για εναλλασσόμενο ρεύμα. Τώρα στην Ενεργειακή Ένωση ε, ακούμε ότι έχει σημασία η περιφερειακή συνεργασία. Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς ενέργειας ανέκαθεν συνεργάζονταν και βελτιώνουμε και εμείς τον συντονισμό μας για να εξασφαλίσουμε τα συστήματα με πολύ μεγάλη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Όπως γνωρίζετε αυτό είναι μεγάλη πρόκληση και θα πρέπει να την απαντήσουμε. Και έχουμε και κέντρα τοπικού συντονισμού και περιφερειακού το 2015 θα συμφωνήσουμε και όλοι οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς θα ε, συγκεντρωθούν. Αναλύουμε θέματα ασφαλείας, χωρητικότητας και άλλα σχετικά. Ολοκληρώνεται, λέει ο Πρόεδρος. Λοιπόν, εργαζόμαστε σε περιφέρειες, όπως είπαμε, και ελπίζουμε όταν θα φτάσουμε στους στόχους του 2030 αυτές οι απαιτήσει του περιφερειακού ε, σχεδιασμού και το ενεργειακό μείγμα να έχει γίνει πραγματικότητα. Είναι για μας προτεραιότητα, είναι για μας πρόκληση και πολύ σημαντική για το μέλλον. Η Ενεργειακή Ένωση έχει δημιουργηθεί για να λύσει αυτό το τρίλημα που σας είπα προηγουμένως, ο σχεδιασμός της αγοράς και η ρύθμιση κυρίως έχουν ολοκληρωθεί και έχει έρθει η ώρα της υλοποίησης. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ε, Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Χάγκεμ. Ο κύριος Μπουζάτση, ο Γενικός Διευθυντής για τα θέματα του αερίου της ΕΝΣΟ. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. ευχαριστούμε για τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε εδώ τη δουλειά της ΕΝΖΟ και να δώσουμε και κάποιες προοπτικές ενιακής ένωσης. Θα σας δώσω μία εικόνα. 26 χώρες από τις 28 Μάλτα και Κύπρος δεν συμμετέχουν ακόμα καθότι δεν υπάρχει σύστημα αερίου στις χώρες αυτές. Έχουμε 242.000 χιλιόμετρα αγωγών για να μεταφέρουμε το αέριο στα διάφορα μέρη της Ευρώπης. 23 περίπου της 100 καλύπτει του ενεργειακού μείγματος, το φυσικό αέριο. Εδώ έχουμε τις διαστάσεις ε, φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού. Σημειώσετε το εξή σημαντικό, το φυσικό αέριο δεν ήταν εκτός της δεκαετίας 50 και 60 όπου είχαμε εθνικές αγορές φυσικού αερίου, από τότε δεν είναι θέμα εθνικής αγοράς αλλά διεθνούς Αγορά όπου οι, ραές, ροές του αερίου περνούσαν από διάφορε χώρε προκειμένου να διοργανώνεται η διανομή και η τελική προορισμή της μεταφοράς. Για τον λόγο αυτό το φυσικό αέριο πάντα υπήρξε ευρωπαϊκή επιχείρηση με όλους τους μεταφορείς στην Ευρώπη. Να θυμίσω ότι οι εισαγωγέ από τη Ρωσία από τις κάτω χώρες και από την Βόρεια Αφρική από τη δεκαετία του 70 και μετά 80 και 90 και τελικά είχαμε από τη Βόρεια Θάλασσα στα τέλη του δεκαετίας του 90. Λοιπόν, ο ρόλος του ENSO-G είναι αντίστοιχος με το ENSO-E. Ομαδοποιούμε λοιπόν τους ε, διαχειριστές μεταφοράς ώστε να προαγάγουμε την, ε, και να υποστηρίξουμε την ε, οργάνωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Να σας δώσω μια ιδέα για την ε, διοικητική δομή. Όλα τα μέλη εκπροσωπούνται το, στη Γενική Ολομέλεια και έχουμε εδώ το Διοικητικό Συμβούλιο με δύο επίπεδα λήψεων αποφάσεων και η δομή που βλέπετε είναι η επιχειρησιακή δομή που ενέχει πάρα πολλά άτομα προκειμένου να έχουμε επιτυχία στα παραδοτέα τα οποία είναι το πανευρωπαϊκό δίκτυο ε, τη, η αξιολόγηση αν θέλετε ε, προσφοράς και ζήτηση αερίου κοινά επιχειρησιακά εργαλεία για την ε, συνεργασία των δικτύων όπως και τα συστήματα δεδομένων και πληροφοριών. Ζητώ συγγνώμη λέει ο μιλητής. Προσπαθώ να ελέγξω τις διαφάνειες. So, ε, Άρα λοιπόν, ε, μία από τις πιο σημαντικές θεματικές για την SOG είναι μια δωδεκάμινη περίοδος προκειμένου να αναπτύσσονται τα έγγραφα, όταν έχουμε λάβει βεβαίως τέτοια εντολή η κλίση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από τα πιο σημαντικά πράγματα στην προετοιμασία του κώδικα του δικτύου είναι η σημαντική συμμετοχή των ενδιαφερομένων φορέων σε όλη την Ευρώπη. Και έχουμε τον τρίτο πυλώνα ας πούμε στην πράσινη περιοχή ε, που είναι μια κοινή επιτροπή όλων των ενδιαφερομένων φορέων ώστε να αναπτύσσεται μια συνένεση, μια συμφωνία επί της προτάσεως που έχει υποβάλει η NSOG. Επομένως η δομή αν θέλετε μαζί με τις ε, κεντρικές ομάδες των Βρυξελών που είναι ο ολιγομελείς υποστηρίζεται απολύτως από το σύνολο των μελών της NSOG με όλους τους ενδιαφερομένους φορείς ώστε να επιτύχουμε στο μέτρο του δυνατού συνένεση επί των προτάσεων. Η συνεργασία φυσικά είναι κεντρική σημασία για την επιτυχία για την επίτευξη οποιοδήποτε στόχου, ιδιαίτερα στα ενεργειακά θέματα, όπου οι ενδιαφερόμενοι φορεί θα πρέπει να ενημερώνονται καταλήλου καθ' όλη τη διάρκεια τη διαδικασία. Και αυτό που έχουμε καταφέρει να συστήσουμε είναι μια ευρεία πραγματικά συμμετοχή προκειμένου να επιτύχουμε τα αποτελέσματα. Και ποια ήταν τα αποτελέσματα. Να έχουμε μια πραγματική εσωτερική αγορά, προκειμένου να την έχουμε, χρειαζόμαστε εργαλεία και κανόνες. Οι κανόνες είναι οι κώδικες του δικτύου και τα εργαλεία είναι τα δεκαετή ε, εφαρμοστικά προγράμματα που δίδουν στην αγορά όλες τις πληροφορίες και εκείνες που χρειάζεται για να λειτουργεί να αγοράζει και να διαθέτει ε, φυσικό αέριο σε όλη την Ευρώπη. Ποια είναι η κατάσταση των ε, κωδίκων δικτύου. Σε αυτά τα τελευταία πέντε χρόνια αυτό που καταφέραμε να προτείνουμε και να εγκριθεί τελικά από την Επιτροπή Φυσικού Αερίου, τρεις κώδικες σχετικά με την ισχύ ή την χωρητικότητα, την ε, εξισορρόπηση που θα εφαρμοστεί από 1η Νοεμβρίου φέτος και 1η Οκτωβρίου αντίστοιχα, θα έχουμε την ε, ε, διαλειτουργικότητα που είχε εγκριθεί από την Κομισιόν 30 Απριλίου και εργαζόμαστε επί της ε, κοστολόγησης και της χωρητικότητος. Σχετικά τώρα με τη διαχείριση των συμφορήσεων, είχαμε μια κατευθυντήρια γραμμή που τελικά ενεκρίθηκε από την Επιτροπή Φυσικού Αερίου Επομένως το συνολικό πλαίσιο υφίσταται, αυτό που λείπει είναι το πιο σημαντικό βήμα που είναι η εφαρμογή τελικώς. Η ένθο G και τα μέλη της όχι μόνο έχουν προετοιμάσει όλα τα έγγραφα αλλά έχουν προχωρήσει και σε δοκιμές και ελέγχους για την ε, πρώιμη εφαρμογή των κωδίκων αυτών όπου οι μεταφορείς ομαδοποιούνται προκειμένου να αναπτύξουν την λεγόμενη πλατφόρμα ε, χωρητικότητος ώστε να δώσουν στους διαχειριστές δικτύου τη δυνατότητα να κρατήσουν συγκεκριμένες ροές στο κάθε βραχαίρο του δικτύου. Επίσης έχουμε εργαλεία μέσω των οποίων η αγορά λαμβάνει πληροφορίες επί τη βάση μιας ενιαίας πλατφόρμας για την διαθεσιμότητα και τη χωρητικότητα παντού. Έτσι λοιπόν κάθε τελικός χρήστης έχει μία εικόνα ασφαλής σχετικά με το πού μπορεί να μεταφέρει το αέριό του και πόσο μπορεί. Η διαφοροποίηση τώρα είναι πολύ σημαντική για την ε, ανάπτυξη της ε, αγοράς ενέργειας και προκειμένου να διαφοροποιήσουμε λοιπόν τις οδούς ε, εφοδιασμού χρειαζόμαστε επενδύσεις. Και γιατί χρειαζόμαστε επενδύσεις και όραμα και, πληροφο... και ενημέρωση και πληροφορίες αν θέλετε. Χρειαζόμαστε επενδύσεις διότι όπως γνωρίζετε η διαθεσιμότητα του φυσικού αερίου στην Ευρώπη κατέρχεται, περιορίζεται στην Ευρώπη και ακόμα και αν ε, εφαρμόσει κανείς τα, τα σενάρια εργασίας, ε, τις υποθέσεις εργασίας και τις προβλέψεις που υφίστανται για σταδιακή μείωση, αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση κατά την οποία συνολικά η εθνική παραγωγή κατέρχεται και επομένως πρέπει να συνδυάσουμε αυτή τη μείωση με άλλες ροές αερίου, βιομεθανείο ή σχιστολιθικού αερίου ή άλλες οδούς μέσα των οποίων θα μπορούσε να εισαχθεί, να εισρεύσει ε, φυσικό αέριο ώστε να είναι βιώσιμη η αγορά. Διαφοροποίηση δηλαδή για να μην είμαστε μόνο με κάποιους προμηθευτές και επομένω με λιγότερες δυνατότητες αν θέλετε ανταγωνιστική ε, εξισορρόπηση στην αγορά. Τώρα όταν μιλούμε για τον εξοπλισμό και τι υποδομέ, μιλούμε για το πώ πρέπει να αναπτύσσονται αυτέ οι υποδομέ και από το δεκαετέ ε, αναπτυξιακό σχέδιο που ενεκρίθη τον τελευταίο μήνα βλέπετε ότι υπάρχουν πάρα πολλά έργα που υποβάλλονται, μερικά έχουν ήδη εγκριθεί, μερικά εκκρεμούν, εκκρεμεί η έγκρισή τους, από τη στιγμή που εγκρίνεται ένα έργο, Are you moving itself? Uh, okay, thank you very much. It's better. I was saying that. Uh, Έλεγα λοιπόν από τη στιγμή που λαμβάνεται η τελική επενδυτική απόφαση μέχρι το να έχει κανείς διαθέσιμο τον αγωγό ή την υποδομή παρέρχεται ένα σημαντικό διάστημα και όπως βλέπετε ε, παραμένουν αρκετά προβλήματα για τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών ή στην Ευρώπη. Και μπορούμε να πάμε στην τελική διαφάνεια από αυτή τη χαρτογράφηση έχετε μια εικόνα της υποδομής που ακόμα είναι απαραίτητη. Η Ευρώπη ούτως ή άλλως χρειάζεται φυσικό αέριο και πρέπει να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα των συστημάτων φυσικού αερίου. Επίσης είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν το συντομότερο δυνατόν όλοι οι κανόνες που έχουμε ήδη στη διάθεσή μας. Ζητώ συγγνώμη αν μακρηγόρησα. Ε, Ευχαριστούμε κύριε Μουζάτσι και κυρία Χάρτιν για την ε, παρουσίαση σας. Κανένας δεν ε, ζήτησε το λόγο από τους συντονιστές. Ε, δεν ξέρω, υπάρχει κάποιος συντονιστής που θέλει το λόγο. Τρία λεπτά καταρχήν και αυτοί που δεν είναι συντονιστές θα έχουν το λόγο για ένα λεπτό. Συντονιστές τρία λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλές πληροφορίες λάβαμε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Με ε, βάση τα blog που παρουσιάσετε από πλευρά ε, προσφοράς ή εφοδιασμού είπατε ότι υπάρχει μείωση παραγωγής. Κατά την άποψή σας το σχιστολιθικό αέριο πόσο σημαντικό θα γίνει και ε, ποια ποσοστιαία αναλογία θα μπορούσε να κατέχει στο μέλλον. το σχιστολιθικό αέριο έχει ένα ρόλο να διαδραματίσει. Ε, έχουμε διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες από τον ΙΠΑ και στην ανακοίνωση για την ενέργεια είπαμε ότι το σχιστολιθικό μπορεί να ευεργετήσει την Ευρώπη. Η χρήση του θα είναι ευεργετική. Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να αποφασίσει για την χρήση του σχιστολιθικού. Τώρα ως προς την ποσοστή αναλογία, δεν θυμάμαι τα αριθμητικά στοιχεία, μπορείτε να τα βρείτε στις διαφάνειες, αλλά και στην ιστοσελίδα μας στο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύων. Για να σας δώσω μια τάξη μεγέθους, το 2020 εν δυνάμει θα έχουμε ένα δις ε, κυβικά μέτρα, αλλά το 2030 οι προβλέψεις που θα πρέπει να επιβεβαιωθούν μπορούν να μας οδηγήσουν σε 20 με 30 δις κυβικά μέτρα που είναι το 1 δέκατον της συνολικής χρήσης. Είχαμε 400 ε, ε, εκατομμύρια πέρσι. Βεβαίως είναι και θέμα περιβάλλοντος και τα κράτη-μέλη θα αποφασίσουν την καλύτερη δυνατή πολιτική. Ξέχασα να πω πριν, επειδή δεν είχα χρόνο, ότι η συνεργασία μεταξύ όλων ήταν το κλειδί κατά την πενταετή συνεργασία του ΕΝΣΟΚ για να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε το δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύων με τη νέα, στη νέα έκδοσή του και έχοντας ε, όλες τις πληροφορίες από τα θεσμικά όργανα και από την Acer, αν θέλουμε να συνεχίσουμε. Διαφορετικά, αν ο καθένας θέλει να ε, δουλέψει μόνος του, τότε θα φτάσουμε στο στόχο. Νίμπλε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για τις ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις σας. Έχω δύο ερωτήσεις το τρίτο ε, πακέτο για την εσωτερική αγορά ενέργειας, αν θυμάμαι καλά. Α, δεν ε, ακούτε, χρειάζεται διερμηνία. Θα το ξαναπώ από την αρχή. Gut, dann ich einfach nochmal Θα ξαναπώ από την αρχή. Σας ευχαριστώ πολύ για τις παρουσιάσεις. Τώρα μπορώ να μιλήσω γερμανικά, ωραία. Έλεγα λοιπόν ότι είχα δύο ερωτήσεις. Αν θυμάμαι καλά, το τρίτο ενεργειακό πακέτο είναι από το 2009, έτσι δεν είναι. Και ισχύει, έπρεπε να είχε εφαρμοστεί μέχρι το 2011 και τώρα έχουμε 2015. Και μιλάμε για μια εσωτερική αγορά ενέργειας και απέχουμε πόρο από αυτή. Αφού έχετε και συμβουλευτικό ρόλο και συμβουλεύετε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι μπορούμε να κάνουμε ακόμα έτσι ώστε να δημιουργήσουμε ε, μια εσωτερική αγορά ενέργειας, να επιταχύνουμε τη διαδικασία. Ακούω ότι έργα γίνονται και πώς τρέχουν, αλλά αν δούμε πόσο επίπονη είναι αυτή η διαδικασία για να εφαρμοστεί ε, σε κάποια κράτη-μέλη, Έχω απογοητευτεί πλήρω. Δεν είναι νέα η κατάσταση. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε την εσωτερική αγορά και ακόμα απέχουμε πάρα πολύ. Εσείς λοιπόν που συμβουλεύετε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι τους λέτε και των κρατών μελών. Και θέλω να σα ρωτήσω προσωπικά για τις αγορές που δημιουργείτε, για τη χωρητικότητα. Στη Γερμανία που είναι η πατρίδα μου κάνουμε και εμείς αυτή τη συζήτηση. Πώς βλέπετε ε, αυτές τις ε, νέες αγορές που χτίζεται και την χωρητικότητα. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Um, the speed. Το θέμα της ταχύτητας είναι πολύ σημαντικό. Στην πατρίδα μου λέω ότι δεν τα καταφέραμε με τα δύο πρώτα ε, πακέτα, αλλά το τρίτο είναι τόσο λεπτομερές, ενέχει πολλούς κανονισμούς και θα πρέπει να το εφαρμόσουμε το ταχύτερο δυνατόν και βέβαια θα πρέπει να υπάρχει η ενιαία αγορά, οι κανόνες υπάρχουν, έχουμε εντάξει όλα τα στοιχεία, ακόμα και τα εθελούσια στοιχεία και όλα είναι έτοιμα. Τώρα ως προς την ε, ταχύτητα θα πρέπει οι διαχειριστές δικτύου να το ε, δουν αυτό το θέμα και να το εφαρμόσουν το συντομότερο δυνατόν. Το Acer θα πρέπει να έχει όλα τα μέσα στη διάθεσή του για να μπορέσει να εφαρμόσει αυτό το πλαίσιο. Ο κανονισμός υπάρχει. Ίσως υπάρχουν ορισμένα στοιχεία που λείπουν όπως η ασφάλεια προμηθείων, η ασφάλεια φοδιασμού, ορισμένοι κανονισμοί, η σύνδεση λιανικής αγοράς και χονδρικής, αλλά όταν το πακέτο ε, εγκριθεί, δηλαδή οι κώδικες δικτύου, τότε θα έχουμε όλα τα στοιχεία, αλλά θα πρέπει να δούμε πρώτα την εφαρμογή και όλοι θα πρέπει να συμμετέχουμε ενεργά. Υπάρχουν τα μέσα και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ασκήσουν πίεση. Είμαι αρκετά αισιόδοξη ως προς την αγορά χωρητικότητας, ως προς τη χωρητικότητα στο ένσο λέμε ότι θα πρέπει να ορίσουμε ένα πρότυπο στόχων, δηλαδή να έχουμε μία ενιαία ενεργειακή αγορά και όχι να μπούμε σε θέματα χωρητικότητας αν δεν δούμε πριν την αγορά ενέργειας. Μπορούμε να έχουμε καλύτερο χρονισμό, μπορούμε να βγάλουμε την ευελιξία, μπορούμε να επιταχύνουμε και να μην ε, περιμένουμε με σταυρωμένα χέρια και μετά να εφαρμόσουμε την αγορά για τη χωρητικότητα. Δηλαδή πρέπει να έχουμε μία ενιαία αγορά ενέργειας καταρχήν και μετά να δούμε και τα θέματα της χωρητικότητας στη συνέχεια. Όχι σε εθνικό επίπεδο αλλά σε ευρωπαϊκό. Και θα πρέπει να έχουμε και μία διασυνοριακή διάσταση. Δεν θα πρέπει να σταθούμε στα εθνικά σύνορα εφοδιασμού γιατί θα είναι πολύ δαπανηρό το σύστημα. Αλλά καταρχήν η ενέργεια. Ο κύριος ε, Κέλλη. Ευχαριστώ πολύ και για τις παρουσιάσεις και τη συνεισφορά σας. Δύο ερωτήσει μόνο έχω. Ε, μία ερώτηση για τον καθένα. Μήπω να τα λέτε πιο κοντά στο μικρόφωνο. Ναι, δύο ερωτήσει έλεγα. Μία για τον καθένα. Πρώτη. Για τις απαιτούμενες επενδύσεις μέχρι το 2030. Ε, μιλήσατε για το 150 δις. Πού θα τα βρείτε και θα τα βρείτε και αν όχι ποιες θα είναι οι συνέπειες. Γενικά για το φυσικό αέριο πριν από λίγες εβδομάδες είχα την ευκαιρία και τη χαρά να μιλήσω σε μια διάσκεψη στην Ιρλανδία εκεί στο Δουβλίνο γιατί η γεωπολιτική κατάσταση Ουκρανία-Ρωσία μας αφύπνισε στην Ευρώπη και μας έκανε να ψάχνουμε διαφοροποίηση ε, των πηγών. Το υγροποιημένο φυσικό αέριο νομίζω είναι μια αγορά ε, για μας που ανοίγει και είναι καλό γιατί υπάρχουν και άλλοι προμηθευτές. Τι γίνεται με το ε, βιολογικό, το βιοαέριο. υπάρχει χώρο στην αγορά και θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Δηλαδή είναι ανταγωνιστικό αυτό το προϊόν σε σχέση με το φυσικό αέριο και ε, το υγροποιημένο. Απαντήσετε για τα επενδυτικά. 150 δισεκατομμύρια ευρώ είναι ο σχεδιασμός μέχρι το 2030 και θα προέλθουν αυτά τα χρήματα από τους πελάτες του δικτύου. Είναι τεράστια τα ωφέλη και πιάνουν τόπο οι επενδύσει. Επενδύει ένα ευρώ και σου αποδίδει δύο. Είναι πολύ κερδοφόρα επένδυση. Αν είχα χρήματα, εγώ εκεί θα επένδυα. Είναι καλό αυτό λοιπόν ε, η προοπτική. Θέλουμε ένα σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο, αυτό χρειαζόμαστε, έτσι ώστε να αποδίδει η επένδυση με τρόπο αποδεκτό και στις περισσότερες χώρες αυτό ισχύει ήδη, διότι το βλέπουν και τα κράτη-μέλη και κατανοούν πόσο σημαντικό είναι να οικοδομούν αυτά, να χτίσουν τα δίκτυα. Τα χρήματα είναι πάντα πρόβλημα ε, βρεθούν, αλλά ε, αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρχει ένα σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο και είναι θετικά τα όσα βλέπουμε αυτές τις μέρες perspective you said about... Υπό την οπτική γωνία του φυσικού αερίου αναφερθήκατε στην Ρωσία και την Ουκρανία και τα προβλήματα που θα μπορούσαμε να έχουμε με τον εφοδιασμό. Προφανώς πρέπει να το λάβει κανείς αυτό υπόψη του προκειμένου να επενδύσει στις διάφορες μορφές αερίου το υγροποιημένο, το βιοκαύσιμο και για άλλες εναλλακτικές λύσεις αερίου. Το βιοαέριο δεν ανήκει στα εναλλακτικά, αλλά εν πάση περιπτώσει εφόσον υπάρχει αποδεκτή ποιότητα, κανονικά δεν προβλέπουμε άλλα προβλήματα. Τώρα, οι επενδύσεις είναι πάντα εξαιρετικά σημαντικές. Προκειμένου να έχει κανείς μια πραγματική εσωτερική αγορά. Όπως έλεγα και πριν, χρειαζόμαστε τους κανόνες, το πλαίσιο των κανόνων και τους έχουμε για το φυσικό αέριο. Μετά πρέπει να τους εφαρμόσουμε, το οποίο σημαίνει όλοι από κοινού, με κοινή ευθύνη, όπου ο καθένας θα αναλαμβάνει το μερίδιο που το αναλογεί της ευθύνης αυτής. Μετά θα πρέπει να δουλέψουμε μεταξύ των ε, δικτύων μεταφορών των ε, αρχών, των κρατών μελών και σε περιφερειακό επίπεδο ενδεχομένω, προκειμένου να βελτιστοποιήσουμε την κατάσταση των διασυνδέσεων που είναι απαραίτητες για να ξεπεράσουμε κάποια κενά που έχουμε σε προβλήματα. Αναφέρομαι στην περιοχή της Βαλτικής και σε κάποιες περιοχές της Ανατολικής Ευρώπης λόγω ακριβώς κατάστασης ε, με τη Ρωσία. Επίσης χρειάζεται σταθερότητα ρυθμιστικού πλαισίου Θυμίζω ότι στι ΗΠΑ υπάρχουν σταθεροί ρυθμιστικοί κανόνες τα τελευταία 10 χρόνια και πλέον. Αυτό απαιτείται προκειμένου να προσελκύσει κάποιος τους επενδυτές. Γιατί κάποιοι ρωτήσατε ποιος θα βάλει τα χρήματα. Και η Μπέντε είπε ότι και ο επενδυτής πρέπει να καταλάβει ότι αξίζει τον κόπο να επενδύσει στο φυσικό αέριο ή στον ηλεκτρισμό. Το οποίο σημαίνει, ιδιαίτερα για το αέριο, ότι πρέπει κανείς να έχει ένα, ένα όραμα σχετικά με το ενεργειακό μείγμα. Ιδάλλως δεν μπορούμε να βρούμε τον επενδυτή, όχι εκείνον που θα κατασκευάσει μόνο την υποδομή, αλλά που θα επενδύσει στο πεδίο του φυσικού, στην αγορά του φυσικού αερίου. Είτε μιλούμε για LNG, είτε μιλούμε για βιοαέριο, είτε οτιδήποτε άλλο. Για να το μεταφέρει από την μονάδα επεξεργασίας υγροποίησης μέχρι το δίκτυο διανομής. Και ε, υπάρχουν και αρκετές λύσεις που αναπτύσσονται τοπικά. Από τη στιγμή όμως που διοχετεύεται το αέριο στο δίκτυο δεν μπορεί να σφαραγίζει κανείς τα μόρια του γιατί είναι στο σύστημα πλέον η δική μου αίσθηση είναι ότι το βιοαέριο θα, θα συμβάλλει μάλλον σε τοπικό επίπεδο. Εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία γιατί από τη στιγμή που όπως έλεγα θα μπει στο δίκτυο θα συμμετέχει στο μείγμα. Χρειάζεται λοιπόν σταθερότητα ρυθμιστικού πλαισίου, χρειάζεται κίνητρα για τους επενδυτές, να έχουμε ένα όραμα για το ενεργειακό μείγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το φυσικό αέριο, για την ηλεκτρική ενέργεια και για κάθε άλλη ενεργειακή πηγή. Ο Πρόεδρος. Και εγώ θα ήθελα να σας υποβάλω μια ερώτηση μαζί με τους συναδέλφους, ε, κύριε Μουζάτση, σχετικά με την, ε, μετά της εφαρμογής. Βλέπω μια λευκή κοιλίδα στην Ελβετία, δεν βλέπω και την Ευρωβηγία λέει ο πρόεδρος κοιτώντα την κυρία Χάγκεμ. Και δεν βλέπω και τη Φιλανδία και τη Σουηδία. Εσείς μπορείτε να μου το εξηγήσετε. Αν θυμόσαστε το χάρτη της ε, Ευρώπης ε, για την ΕΝΣΟΚ, βλέπετε ότι η Ελβετία είναι μέλος μας και η Νορβηγία, η Ουκρανία, έχουμε και την Ουκρανία και την Φύρομ. θα δούμε κατά πόσο υπάρχει και άλλων ενδιαφέρον και θα προωθήσουμε συνεργασία και με άλλες χώρες. Η Ελβετία δεν είναι στο χάρτη γιατί δεν είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γι' αυτό υπάρχει αυτή η κοιλίδα, η λευκή κοιλίδα. Η Σουηδία δεν εμπεριέχεται γιατί δεν ξέρει σε ποια πλατφόρμα θα συμφωνήσει. Εδώ έχετε την πλατφόρμα χωρητικότητας μπροστά σας και δεν έχει προσχωρήσει σε μία από τις τρεις πλατφόρμες η Σουηδία. Όπως είπα και πριν, καλύπτουμε οι 26 από τα 28 κράτη-μέλη και τέσσερις χώρες, ε, Ελβετία, Νορβηγία, Φύρον και Ουκρανία. Άλλες ερωτήσεις παρακαλώ προς τους ε, προσκαλεσμένους μας. Όχι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κύριοι ε, Μουζάτσι και Χάγκεν, για τη συμμετοχή σας στη συζήτηση. Και τώρα φτάνουμε στο τελευταίο θέμα της ε, σημερινής συνάντησης. Όπως ξέρετε έγινε μια αποστολή στην Ουάσιγκτον και την Πενσιλβανία και ήρθαμε σε επαφή με μέλη του Κογκρέσου που αυτή τη στιγμή επισκέπτονται τις Βρυξέλλες και ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση μαζί τους. Εδώ είχαμε, έχουμε μάλλον μέλη που συμμετείχαν σε αυτή την αντιπροσωπεία, στην αποστολή αυτή και θα θέλαμε να μας ενημερώσετε. Ίσως ο κύριος Ρούμπιχ καταρχήν ή ο κύριος Πέτερσον που ήταν ο επικεφαλής. Ο κύριος Πέτερσον θα αρχίσει και ίσως και άλλα μέλη θα μπορούσαν να μας διαφωτίσουν στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Εννέα ε, μέλη της Επιτροπής μας μετέβησαν στην Ουάσιγκτον και την Πενσιλβανία 16 με 19 Μαρτίου 2015 Στη Μεσυλβανία θέλαμε να μελετήσουμε το, στο λιθικό αέριο και στο Οχάιο που τρέχει με ραγδαίους ρυθμούς η παραγωγή. Είχαμε επαφές με εταιρείε παραγωγής ενέργειας, ΜΚΟ, πολίτες, ε, ρυθμιστές ε, και πήγαμε και στο Οχάιο επιτόπου σε μια γεώτρηση. και ε, συναντηθήκαμε και με το τμήμα το τοπικό για την προστασία περιβάλλοντος ε, και ε, ρωτήσαμε αν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των διαφόρων πολιτιών για να προσελκύσουν τις επενδύσεις στο σχιστολιστικό γιατί τα περιβαλλοντικά δεδομένα και πρότυπα δεν είναι παντού τα ίδια. Και ρωτήσαμε τι ισχύει σε επίπεδο ομοσπονδίας και τι ισχύει σε επίπεδο πολιτείας και αν συγκρούεται η δραστηριότητα υδρορογμάτωσης με τη γεωργία ή με άλλες δραστηριότητες οικονομικές και τι ε, διδάγματα εξήφθησαν για την ομοθέσια; Είδαμε και στην νότιο-ανατολική Σιλβανία ε, εκπροσώπους περιβαλλοντικών έργων και θεμάτων δημόσιας υγείας ε, τι γίνεται με την άγρια πανίδα, τα προστατευόμενα είδη και εν γέννη την ε, ε, επίδραση στην ε, δημόσια υγεία. Μας είπε ένας καθηγητής τα δεδομένα, τα επιστημονικά και πόσο επηρεάζει την οικονομία της Πενσιλβανία και του Πίτσμπουργκ. Πήγαμε και στο Οχάιο, στα 120 χιλιόμετρα δυτικά του Πίτσμπουργκ Περάσαμε πολύ ε, ώρα σε λεωφορεία. Η Total εκεί έχει με την Chesapeake ε, ένα ε, joint venture, μια κοινοπραξία και βγάζουν ε, σχιστολιτικό αέριο με συμπίεση και με υδρορογμάτωση και ήταν πολύ ενδιαφέρουσα επίσκεψη εκεί επί τόπου. Στην Ουάσιγκτον συναντηθήκαμε με εκπροσώπους Think Tank, με εκπροσώπους ε, του ε, Υπουργείου ε, Ενέργειας με εκπροσώπους τηλεπικοινωνίας για την ενεργειακή ασφάλεια, Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Ίδρυμα και για τη Διεθνή Ειρήνη για να συναντηθούμε με διαφόρους εμπειρογνώμονες σε θέματα ασφάλειας ενεργειακής Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών είδαμε και μέλη του Κογκρέσου. Και βασικά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πώς να μειώσουμε την εξάρτησή μας από το ρωσικό φυσικό αέριο. Ανταλλάξαμε απόψει με ομολόγους μας ε, της Βολής των Αντιπροσώπων για την ενεργειακή ασφάλεια ε, και ε, το Μάιο τους φιλοξενούμε εδώ εχθές ήρθανε ο Μάικλ Μακόλ, γερουσιαστή, είναι πρόοδο τη Επιτροπή για την Εσωτερική Ασφάλεια και μέλος της Επιτροπή για την Επιστήμη και την Τεχνολογία και μιλήσαμε για ε, υψηλή τεχνολογία, μεταφορά τεχνογνωσίας και ενεργειακό εφοδιασμό. Στο Υπουργείο Ενέργειας συναντηθήκαμε με τον κύριο Κρίστοφερ Σμιθ που είναι αρμόδιος υφυπουργός για ορυκτά καύσιμα ε, και ήταν και ο κύριος Νίκολας Σέρμαν ο οποίος είναι ο συντονιστής του Συμβουλίου ε, Ενέργειας Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών και αρμόδιος εκεί. Ήταν από τις καλύτερες ίσως συνεδριάσεις και επαφές που είχαμε κατά τη διάρκεια όλης της αποστολής ε, ε, Βέβαια ε, συζητήσαμε την έρευνα για το σχιστολιθικό, ε, για νέες τεχνολογίες που θα προστατεύουν τα υπόγεια ύδατα και το περιβάλλον. Έχει διαπιστωθεί ότι έχουν αυξηθεί οι σεισμοί στις περιοχές που γίνεται τέτοια εξόριξη. Συναντηθήκαμε και με την Επιτροπή, Ομοσπονδιακή Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών για το διαδίκτυο και τη σχετική νομοθεσία που πρόσφατα εγκρίνανε. Ε, ολοκληρώνοντας, Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους For such a good and interest. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η αποστολή, αντιπροσωπεία. Ε, είχαμε πάρα πολύ γόνιμες συζητήσεις με τους Αμερικανούς ομολόγους μας. Ήταν μεγάλη ευχαρίστηση η ε, συμμετοχή. Ευχαριστώ και τη γραμματεία. Ήταν τεράστια η ε, ε, προετοιμασία και ακόμα μεγαλύτερη υπομονή που έδειξαν προς τα μέλη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. αυτή πολύ ενδιαφέρουσα σύνοψη της επίσκεψής σας καθότι την έχετε και γραπτός ε, και έχουμε και πολλούς απόντες ε, θα μπορούσαμε μήπως να την επισυνάψουμε ε, στα πρακτικά τη σημερινή συνεδρίαση για να μπορούν και άλλοι συνάδελφοι να τη δουν γιατί ξέρουμε ότι 12 μέλη είχαν συμμετάσχει και καλό θα ήταν να δούμε τα συμπεράσματα. Λοιπόν, τώρα ο κύριος ε, Ρούμπης. Ε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ και τη γραμματεία και τον επικεφαλής αντιπροσωπείας μας διότι ο επικεφαλής πραγματικά το οργάνωσε πάρα πολύ καλά, ήταν πολύ προετοιμασμένος και διεύθυνε πολύ καλά τις συζητήσεις. Για μένα δύο είναι τα θέματα που έχουν τεράστια σημασία. Πρώτον, η συζήτηση για το σχιστολιθικό αέριο με τις ΜΚΟ και τις αρμόδιες περιβαλλοντικές αρχές. Έδειξε ότι η τεχνολογία μετεξελίχθηκε ήδη πάρα πολύ και η ασφάλεια και το περιβάλλον πραγματικά είναι στο επίκεντρο για μας. Ήταν πολύ ευχάριστη αυτή η εμπειρία, είναι πάρα πολύ υπεύθυνη η, όλη η διαδικασία εκεί. από την άλλη είδαμε ότι το σχιστολιθικό αέριο τα τελευταία χρόνια δημιούργησε στην Αμερική σχεδόν ένα εκατομμύριο νέες θέσεις εργασίας και έχουν αυξηθεί τα φορολογικά ε, έσοδα και έχουν φτάσει τα 70 δις ευρώ, λέει ο μιλητής δολάρια μας. 40 δις αναμένεται ε, να είναι τα φορολογικά έσοδα δολάρια μέχρι το 2020. Αυτό ε, θα μπορούσε να βοηθήσει τον προϋπολογισμό μας που θα μπορούσε να καλυφθεί τελείως από τα έσοδα. Για το FCC έχουμε την ε, ε, τάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ψηφιακή ενιαία αγορά. Το συζητήσαμε με την Ομοσπονδιακή Επιτροπή ε, Τηλεπικοινωνιών. Και μας είπαν ότι θέλουν κανόνες παιχνιδιού απλούς που να επιτρέπουν ε, τη λειτουργία της αγοράς, να μην εμποδίζουν τους διάφορους φορείς και μπορούμε να συνεργαστούμε με την αντίστοιχη αυτή Επιτροπή των Ηνωμένων Πολιτειών για να επιτύχουμε κάτι ελπιδοφόρο για το μέλλον. Ήταν πολύ ενδιαφέρον το ταξίδι. Είχαμε την ευκαιρία όλοι μας να αξιολογήσουμε πώς μπορούν στο μέλλον να συνεργαστούν επ' αυτών των θεμάτων Αμερική και Ευρώπη. Κάποια άλλη ερώτηση προς τα μέλη που συμμετείχαν στην αποστολή αυτή. Δεν βλέπω, εγώ όμως θα είχα μία, λέει ο Πρόεδρος. Εχθές όταν συναντηθήκαμε με τα μέλη του Κογκρέσου και συζητήσαμε και το σχιστολιθικό αερίο και άλλα ενεργειακά θέματα, κανείς δεν αναφέρθηκε στην πυρηνική ενέργεια. Και αναρωτιέμαι, γιατί αυτό δεν αναφέρεται στην έκθεση της αποστολής. Δεν συζητήσατε καθόλου τα πυρηνικά θέματα με τους Αμερικανούς. Κοιτάξτε, λέει ο κ. Ε, Πέτερσεν. Δεν ήταν μέρος του προγράμματος της επίσκεψης, τα, τα, τα, η πυρηνική ενέργεια. Εστιαστήκαμε κυρίως ε, στο σχιστολιτικό αέριο. Είδαμε και επιχειρήσεις στο πεδίο, fracking ε, και δίσαμε ε, κύριο, κυρίως έμφαση σε αυτά τα θέματα στην, και όχι στα πυρηνικά. Πήγαμε στο Πίτσμπουργκ και μετά στο Οχάιο και πάντοτε η εστίαση εκτός από τα οργανωτικά θέματα ήταν πάντοτε στο σχιστολιθικό αέριο. Είδαμε και πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, αλλά δεν συζητήσαμε καθόλου για τα θέματα πυρηνική ενέργεια. Μάλιστα, λέει ο Πρόεδρο. Να πάω στο τελευταίο λοιπόν σημείο, το οποίο είναι. Καταρχά, διάφορα. Δεν ξέρω αν κάποιος θέλει να προτείνει κάτι υπό τα διάφορα. Εφόσον δεν είναι έτσι, να σας θυμίσω ότι η επόμενη συνεδρίαση έχουμε στις 28 Μαΐου, 9 με 12.30 και μετά το απόγευμα 2.30 με